Pan Przewodniczący! Good morning, colleagues, please. Καλημέρα, παρακαλώ να πάρετε τις θέσεις σας. Αρχίζει η συνεδρίασή μας. Το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τα συμπεράσματα της συνοπτου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 28-29 Οκτωβρίου και οικονομική διακυβέρνηση. Υποδέχομαι και χαιρετίζω την παρουσία στην αίθουσα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του κ. Χέρμαν Βανομπόγιου και την παρουσία επίσης του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του κ. Χωσέ Μανουέλ Μπαρόσο. Επίσης μεταξύ μας έχουμε τους εκπροσώπους της Βελγικής Προεδρίας και Επιτρόπους. Θα αρχίσει η συνεδρίασή μας με μία ενημέρωση και κατόπιν την ομιλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του κυρίου Βαν Ρομπόι. Περίμενε, Mr. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το, η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης και 29ης Οκτωβρίου εστιάστηκε στην οικονομική διακυβέρνηση Ευρώπης,